πίσω τα ψηφίσματα που έχουμε κρίνει στους ενδιαφερομένους που αναφέρονται στο περιεχόμενο των ψηφισμάτων. Λίγη λοιπόν η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.